και αυτών οι οποίε θα υπογραφούν θα δημοσιευτούν με τα πρακτικά αυτή τη συνεδρίαση. Περνάμε τώρα στην υιοθέτηση της ημερήσια διάταξης σύμφωνα με τη μορφή που έχει. Έχω μόνο μία παράκληση για αλλαγή για την πέμπτη. Η ομάδα των φιλελευθέρων ζητάει η έκθεση Balls για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δημοσίων Λογαριασμών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να φύγει από την ψηφοφορία τη ε, Πέμπτη Έχει τον λόγο λοιπόν η κυρία Μπόουλ. Um, ε- Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ω εισηγήτρια για το θέμα αυτό που είχε προγραμματιστεί για ψηφοφορία την Πέμπτη θέλω να πω το εξή. Είμαστε έτοιμοι να το αναβάλουμε για άλλο μήνα το θέμα, διότι πιστεύουμε ότι τώρα ίσως να μπορέσουμε να φτάσουμε στη συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ποια ήταν η κατάσταση. Τέσσερα κράτη-μέλη, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία, δεν ήταν έτοιμε για κάποια στατιστικά στοιχεία που έπρεπε να υποβληθούν υποχρεωτικά. Αυτό ήταν το αδιέξοδο στο οποίο καταλήξαμε στο τέλος της Δανέζικης Προεδρίας. Υπήρξε μεγάλη κάλυψη από τα ΜΜΕ του θέματος και η νέα Προεδρία κατόρθωσε να ασκήσει κάπως μεγαλύτερη πίεση και υπάρχει ενδεχόμενο προσωρινή συμφωνία. Πρέπει να περιμένω να υποβληθεί, αλλά είναι θέμα επίγον προφανώς, διότι το πώς συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία και κυρίως από περιφέρειες, διότι αυτό αφορά το θέμα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχουν εκπλήξεις στα λογιστικά και όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και για όλα τα σχετικά ζητήματα, θα συμφωνεί μαζί μου το Κοινοβούλιο και όλε οι πολιτικέ ομάδε ότι αυτό είναι σημαντικό. Και θα συμφωνούν με την πρόταση για την αναβολή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι κάποιος υπέρ του αιτήματο. Κατά. Οπότε θα ψηφίσουμε. Όποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές οπότε φεύγει από την ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα οπότε έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη αυτής της εβδομάδας και τώρα ξεκινάει η συζήτηση για το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξη έκθεση της κυρίας Λάρα Κόμη για την ευρωπαϊκή τυποποίηση η κυρία Κόμη λοιπόν έχει τον λόγο η συγκεκριά παρακαλώ